Pan Przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας. Έχουμε μια πολύ σημαντική στιγμή μπροστά μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αύριο θα χαιρετήσουμε την 7η επέτειο μνήμης στα θύματα της τρομοκρατίας, της 11ης Μαρτίου, που είναι αφιερωμένη στα χιλιάδες θύματα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Οι τρομοκράτες έχουν κηρύξει τον πόλεμο κατά των πολιτών χτυπούν σε μέρη όπου κανονικά ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ασφαλής μέσα στη χώρα του. Πρόκειται για μια επονίδιστη, ύπουλη και δειλή συμπεριφορά. Γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει δικαιολογία για την τρομοκρατία. Οι Ευρωπαίοι είναι ενωμένοι και ισχυροί και καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν μπορεί να αποδυναμώσει την πίστη μας και την πεποίθησή μας στις αξίες οι οποίες έχουν χτίσει και ενώνουν την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι όλοι σε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας. Thank you. Ευχαριστώ. Czytam Państwu na początku oświadczenia pisemne. Ξεκινώντας θα ήθελα να κάνω Ορισμένε παρατηρήσει σχετικά με τι ε, γραπτέ δηλώσει που έχουν παρουσιάσει οι συνάδελφοι Μάρκ Ταραμπέλα, Ρετζίνα Μπάστος, Πασκάλ Κάνφιν, Μαρή Κριστίν Βευσιά, Ρενάτ Βέμπερ ως προς τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Καθεστώτος Καταστατικού για την ε, αλληλασφαλιστική εταιρεία, τον συνεταιρισμό και το Ίδρυμα